Good morning. Bonjour. I will in Portuguese. Ξεκινάμε καλημέρα σας, θα συνεχίσω να μιλάω στα πορτογαλικά. Λοιπόν, το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση αυτής της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν προτείνετε κάποιες αλλαγές, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διατάξη. Σημείο 2 είναι οι ανακοινώσει ε, της Προέδρου. Θα λάβατε πληροφορίες που αφορούσαν τις πλέον πρόσφατες ε, ληφθήσεις αποφάσεις. Δεν έχει τίποτα να προσθέσουμε, λοιπόν, στο σημείο 2. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών της 18 Σεπτεμβρίου 2013. Έχετε λάβει και αυτές τις συστάσεις. Οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως εγκεκριμένες από την Επιτροπή. Σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της Δευτέρα Σεπτεμβρίου 2013. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά αυτά, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και μπορούμε να προχωρήσουμε να πάμε στο σημείο 5. Η Σαουδική Αραβία, οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η συντάκτρια από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι η Μπάρμπαρα Ματέρα. Δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα, οπότε η Ρετζίνα Μπάστος θα πάρει το λόγο και θα μιλήσει εκ μέρους της. Έχεις το λόγο. Ναι, ε, λυπάται που δεν μπορεί να παρίσταται η κυρία Ματέρα. Μου ζήτησε λοιπόν να σας περιγράψω κάπως, να σχεγραφίσω το σχέδιο αυτό της γνωμοδότησης και αυτό θα κάνω τώρα. Θα διαβάσω λοιπόν το σημείωμα που μου έστειλε, μου έδωσε. Λοιπόν, η πρόθεση των γυναικείων δικαιωμάτων είναι μία από τις βασικές αρχές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να προωθεί τα δικαιώματα αυτά μόνο εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσης αλλά και στις σχέσεις με τρίτες χώρες. Έχει γεωγραφική σημασία αυτό και στρατηγική σημασία. Η Μέση Ανατολή είναι πολύ σημαντικός χώρος, σημαντική περιοχή, όπου εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις ε, δημιουργούν εμπόδια για τις γυναίκες. Δοθέντος του κενού και το διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, δεν υπάρχει σωστή αντιπροσώπευση των γυναικών στα διάφορα βήματα. Παρουσιάστηκε γνωμοδότηση στη Σαουδική Αραβία σαν μία από τις χώρες όπου εκεί τα δικαιώματα των γυναικών ε, δεν εφαρμόζονται και οι γυναίκες είναι υποδέστες από τους άντρες στα δικαιώματα. Ε, με βάση διάφορα διατάγματα του βασιλιά έγιναν κάποια βήματα για βελτιώσεις. Ε, έχει γίνει πρόσφατη πρόοδος, οι γυναίκες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, αυτή είναι μια βελτίωση, και οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να εκλεγούν στις τοπικές εκλογές το 2015. Και από το 2013, από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και πέρα, οι γυναίκες μπορούσαν να συμμετέχουν σε τοπικά συμβούλια και είχαν δικαίωμα σε αυτό το επίπεδο. Αυτή η βελτίωση είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Ζητάμε από την Ένωση να συνεχίσει το διάλογο με την Σαουδική Αραβία, ούτω ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η ισότητα των φύλων και να βελτιωθεί και το επίπεδο διαβίωσης των γυναικών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή των αρχών της Σαουδικής Αραβίας για το φαινόμενο των καταναγκαστικών γάμων και που γίνεται σε πολύ μικρή ηλικία σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτοί οι γάμοι. Αυτό αντιπροσωπεύει μία παραβίαση της σύμβασης ε, της σχετικής με τα δικαιώματα των παιδιών. Η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες που έχει υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Δοθέντος του ρόλου της, ε, που διαδραματίζει εκεί, γείται το αραβικού κόσμου στην περιοχή. Λοιπόν, για αυτό το λόγο η Σαουδική Αραβία έχει δυνατότητα να παίξει ένα θεμελιώδη ρόλο για την προώθηση της αξιοπρέπειας, της ακαιρεότητας και των δικαιωμάτων των θεμελιωδών των γυναικών. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάστος. Δεν βλέπω κάποιον να έχει ζητήσει το λόγο για το θέμα αυτό και να εκφράσει τοποθετήσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων. θα σας πω ότι έχουμε εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, τον Claude Βερον Plevy, και θα το δώσω αυτό, θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, εκτιμούμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Εκτιμούμε και εμείς αυτά τα περιορισμένα βήματα που έκανε η Σαουδική Αραβία για να δώσει περισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες Σημειώνουμε όπως και εσείς το ότι 30% των γυναικών έχουν διοριστεί ε, σε διάφορους τοπικούς φορείς και η συζήτηση εντοπική ε, για την ε, βία εντός των οικειών, στη οικογενειακή βία συζητείται και αυτό είναι κάτι που είναι πρόσδεκτο. Παρακολουθούμε και τη συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών να οδηγούν. πολλά πρέπει να γίνουν όπως υπογραμμίσατε και θα τονίζουμε αυτά τα σημεία πάντα στις συναντήσεις που θα έχουμε με εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε μαζί μας τον πρεσβευτή του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος και εκείνο έχει ζητήσει το λόγο. Καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά αποτελεί μεγάλη χαρά ε, για μένα που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας. Η ισότητα και τα θέματα ε, που αφορούν τις γυναίκες από το στόμα ενός άντρα. Ε, εντάξει, με φοβίζει λίγο το ότι έχω αναλάβει αυτό το ρόλο εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι παραγωγικός και χρήσιμος. Πρώτα απ' όλα γνωρίζω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο και αυτό δεν βοηθεί, βοηθά και εμένα βέβαια. Δεν μπορώ να καλύψω τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά εξέτασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής σας, καθώς και τις συστάσεις της εισηγήτριας. Πράγματι η Σαουδική Αραβία Ήδη έχει διανύσει πολύ δρόμο ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα και την κατάσταση των γυναικών. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ορισμένα από αυτά ε, για να δείτε ότι ε, η Σαουδική Αραβία τελικά είναι νεαρή χώρα, 83 ετών μόνο. Είμαστε όμως μεταξύ των ιδρυτών των Ηνωμένων Εθνών, είμαστε από τις λίγες χώρες ουσιαστικά οι οποίες έχουν βοηθήσεις και στη σύνταξη της διαρκής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. με βουλευτές, με την άδειά σας θα ήθελα να σας διανύμω και ένα έγγραφο για όλα τα μέλη της Επιτροπής σας σε σχέση με τα μέτρα για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αν θέλετε έτσι, μια υπόμνηση όλων όσων έχουν γίνει και φυσικά ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές σας συστάσεις. Σίγουρα ό,τι σας πω τώρα και ό,τι έγραφε σας διανύμω δεν είναι αρκετά. Εγώ είμαι ο πατέρας τεσσάρων κοριτσιών, να έχετε υπόψη σας, άρα καταλαβαίνω πολύ καλά ε, τα άκρο σεβαστά, δικαι... Ε, τις άκρο σεβαστές διεκδικήσεις και αιτήματα των γυναικών. Ήμουν και μέλος ε, του ε, Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενέβης για δύο θητείες συγκεκριμένα και έχω εργαστεί σκληρά για την πρόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην χώρα μου, Σαουδική Αραβία. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει επίσημη επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα πλέον στη χώρα που ασχολείται άμεσα με τα θέματα αυτά ο βασιλιάς μας είναι αυτός ο οποίος έχει την άμεση αρμοδιότητα. Υπάρχει βέβαια και Εθνική Εταιρεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία ασκεί έντονες πιέσεις σε όλες τις αρχές, ώστε να υπάρχει ισότητα άντρων και γυναικών Νομίζω τα τελευταία δέκα χρόνια ε, έχουμε τέτοιες εξελίξεις που αρχίζουν πλέον οι άντρε Πιστεύω θα αρχίσουν σύντομα να διεκδικούν δικαιώματα, γιατί οι γυναίκες αποκτούν πολλά δικαιώματα στη χώρα Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1961, Τέσσερι ε, ήταν μόνο οι κοπέλες στο σχολείο, τα κορίτσια. Σήμερα έχουμε 6 εκατομμύρια φοιτητές, ε, το 52% εξ αυτών είναι κοπέλες στα πανεπιστήμια έχουμε στην παρούσα φάση αναλογία ένα προς ένα θα έλεγα. 450.000 είναι οι άντρες φοιτητές και οι κοπέλες οι φοιτήτρες είναι γύρω στις 426.000. Σίγουρα και οι γεννήσεις ε, ωφελούν, αν θέλετε, το γεγονός ότι αυξάνεται ο γυναικείος πληθυσμός ε, και σε λίγα χρόνια θα έχουμε 60% γυναίκες στη χώρα μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μελετήσετε τις πληροφορίες που θα σας διανύμω Φυσικά και εγώ προσωπικά και το γραφείο μου, η πρεσβεία μας και η κυβέρνησή μας είναι απόλυτα διατεθειμένη και έτοιμη ε, να έχει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία μαζί σας και να σας παράσχει όλες τις πληροφορίες που θα ζητήσετε. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σας και σας ε, ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ζινοβάστη που εκπροσωπεί την εισηγήτρια. Στο όνομα της κυρίας Μπάρμπαρα Ματέρα επιθυμώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν, ευχαριστώ και τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας που είναι παρόν και αυτό το γεγονός δείχνει ότι υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ισότητας των φύλων. Εμείς ως Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών θα παρακαλέσουμε να συνεχιστούν οι πρόοδοι έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ισότητα των φύλων στην Σαουδική Αραβία. Και θα παρακολουθούμε βεβαίως τα βήματα προόδου που επιτελεί η χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Μία σύντομη παρατήρηση, λέει η Πρόεδρος. Πρώτα θα ήθελα να πω στον εξοχότατο κύριο Πρέζη ότι υπάρχουν και άνδρες μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών που τυχαίνει να μην είναι παρόντες διότι βρίσκονται κάπου αλλού στο Κοινοβούλιο, αλλά η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών δεν σημαίνει ότι τα μέλη είναι μόνο γυναίκες. Έχουμε λοιπόν και άνδρες μέλη. Δεύτερο, Εγώ γνωρίζω τη Σαουδική Αραβία διότι προ 20 ετίας είχα βρεθεί εκεί και ελπίζω ότι υπήρξαν ε, και γνωρίζω ότι υπήρξαν μεγάλες πρόοδοι από τότε διότι τότε προ 20 ετίας δεν υπήρχε απολύτως καμία ισότητα των φίλων στην ε, Σαουδική Αραβία. Είχα υποχρεωθεί τότε να φορώ αυτό το τσαντόρ το οποίο κάλυπτε όλο μου το σώμα και το πρόσωπο μάλιστα τότε δεν επιτρεπόταν καν να εκδοθούν προξενικές θεωρήσεις για τις γυναίκες εγώ μπόρεσα να μεταβώ εκεί διότι συνόδευα τον διπλωμάτη σύζυγό μου κατά κάποιο τρόπο ήμουνα η σκολικοειδής απόφυση του συζύγου μου αν θέλετε να σας το πω έτσι όμως οι αλλοδαπές γυναίκες κανονικά δεν λάμβαναν ε, προξενικές θεωρήσεις και ούτως ή άλλως έπρεπε να συνοδεύονται πάντοτε από άνδρες και δεν επιτρεπόταν να ε, εξέλθουν μόνες τους ε, στους δρόμους. Εξακολουθούν να μην, εξακολουθεί να μην επιτρέπεται να οδηγούν αυτοκίνητο. Γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει ορισμένες πρόοδοι, όχι τόσες πρόοδοι ή τόσο μεγάλες όσο θα θέλαμε να δούμε το γεγονός όμως, εγώ συμφωνώ με την κυρία εδώ, το γεγονός ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ ως πρέσβης της χώρας σας, αυτό δείχνει ότι οι Σαουδάραβες ενδιαφέρονται για το θέμα και ενδιαφέρονται για το τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, για το θέμα της ισότητας των γυναικών. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στα διάφορα μέρη του κόσμου. Ο πρέσβης, με μεγάλη μου χαρά είμαι παρόν εδώ, εξοχότατη κυρία Πρόεδρος. Όπως λένε και στα αγγλικά, seeing is believing. Ελάτε να δείτε με τα μάτια σας, στη Σαουδική Αραβία, οι ίδιες εσείς τι γίνεται την τεράστια εξέλιξη και τις αλλαγές που έχουμε δει εμείς. Έχουμε γυναίκες αναπληρωτές υπουργούς. Έχουμε γυναίκες μέλη των Συμβουλίων Σούρα. Γυναίκες παντού, κυρία Πρόεδρε. Όταν έχετε λοιπόν την ευκαιρία, το γραφείο μου θα σας διευκολύνει για να επισκεφτείτε τη χώρα μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος Εστρέλα. Και συνεχίζει. Αυτή η έκθεση διαθέτει προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών την 8η δεκάτου στις 17 ε, ώρες το απόγευμα. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει στις 26 ενδεκάτου στη ΔΕΝ Επιτροπή Εξωτερικών στις 5 δωδεκάτου. Και στην Ολομέλεια θα καταλήξει μάλλον, του χρόνου. Θα έρθω τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι το υπαριθμό 6. Ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης. Όπου και εδώ συντάχθεια της γνωμοδοτήσεως είναι η κυρία Ματέρα και εν απουσία της η κυρία Μπάστος θα ε, λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας ε, Ματέρα που δεν μπορεί να είναι εδώ για να παρουσιάσει την έκθεσή της. Μου άφησε όμως ένα σημείο που θα διαβάσω. Λοιπόν, τα, τα, τα δικαιώματα γυναικών είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση για την Ευρωπαϊκό Έτος της Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα Όσον αφορά αυτή τη γνωμοδότηση θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει να διατεθούν ευρωπαϊκοί πόροι προς την πρωτοβουλία της ανάπτυξης στις περιοχές του κόσμου που οι γυναίκες είναι αντικείμενα διακριτικής μεταχείρισης. Θυμηθείτε ότι η προστασία της ισότητας των φύλων είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παραδείγματος χάρη η αρχή της ισότητας της αμοιβή συμπεριελήφθη το 1957 στη συνθήκη της Ρώμης εντός των συνόρων της Ενώσεως το πρώτο στάδιο όσον αφορά την απασχόληση, τα πρώτα βήματα για την απασχόληση έχουν επιτευχθεί. Από το 1998 είχαμε αύξηση κατά 8% της απασχόλησης των γυναικών. Εδώ και 15 χρόνια οι μισθωτές γυναίκες, εδώ και 15 χρόνια ήταν 50% του ενεργού πληθυσμού οι γυναίκες. Σήμερα αυτή η αναλογία φτάνει το 60%. Αυτά είναι θερητικά στοιχεία και πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για την εξωτερική δράση όσον αφορά την στήριξη των γυναικών και των κοριτσιών στις τρίτες χώρες. Όλα αυτά στο πλαίσιο του σεβασμού της στρατηγικής για την ισότητα ανδρών και γυναικών για το μέλλον. Έχουν σημασία αυτά τα χρήματα για την ανάπτυξη και αυτά που δίνουν οι δανειοδότες στον κόσμο, οι δωρητές στον κόσμο και θα πρέπει να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα μέσα που εγγυώνονται την επιτυχία της αυτής στις ε, τρίτες χώρες. Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί μόνο παραβίαση των δικαιωμάτων που έχει για την φυσική και ψυχολογική της υγεία, αλλά έχει και αντίκτυπο κοινωνικό και οικονομικό. Χρειάζεται επανεξιολόγηση, πλήρης επαναξιολόγηση του ρόλου των γυναικών στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η προστασία των δικαιωμάτων γυναικών πρέπει να εξεταστεί σε ευρύ πλαίσιο. Χρειάζεται η προστασία των γυναικών στις συγκρούσεις, στους πολέμους και στις ζώνες που αντιμετωπίζουν κρίση. Πρέπει να πρωταγωνιστούν οι γυναίκες στη διαδικασία ειρήνευσης και στην αποκατάσταση της ομαλότητας μετά από συγκρούσεις. Μόνο αν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι γυναίκες μπορούν να παίξουν το ρόλο τους ως επιχειρηματίες και να βρεθούν σε ίση θέση επαγγελματικά με τους άντρες. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο μέσω των διαθεσίμων πόρων να προωθήσουμε τις κάτω πτυχές. Κατάρτιση γυναικών. Αύξηση δυνατότητων απασχόλησης. Να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Κλείνοντας, πιστεύω ότι θα πρέπει να βεστιτοποιηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και να ενισχύσουν συνεχίσουν την προώθηση της ισότητας των φίλων Να παρακινήσουν τις ηγέτες να το κάνουν. Και θα πρέπει να στηριχθεί σε των γυναικών στον κόσμο. Αυτή θα είναι μια απαραίτητη συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φίλων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάστους. Κυρία Παπαδοπούλου. As Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, το 2015 είναι ένα κομβική χρονιά για την ανάπτυξη και είναι και η τελευταία χρονιά για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και για τη λήψη πολύ σημαντικών αποφάσεων για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ορατή. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια από το 1957. Όμως, ναι μεν είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και ιδίως ε, σε τρίτες χώρες, όμως η εξωτερική δράση της Ένωσης δεν είναι τόσο ορατή. Γι' αυτό λοιπόν με τις τροπολογίες μας ε, αποσκοπούμε ε, στο να τονίσουμε τον ρόλο των γυναικών για τη βελτίωση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκε μπορούν να είναι άξονες φορείς αλλαγής και βέβαια μπορούν να, να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στους Ευρωπαίους πολίτες και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους ε, Ανάπτυξης 2015. Δηλαδή με τις τροπολογίες μας θέλουμε να τονίσουμε ότι πρέπει να τονωθεί το ενεργό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και ο ηγετικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την προώθηση της ισότητας των φύλων να είναι σε οι Ευρωπαίοι σε αυτόν τον τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για την αυτοεκτίμηση των γυναικών, τη βελτίωση των γνώσεων που έχουν για τα διάφορα προβλήματα στο τομέα τη υγεία, διάφορες δυνατότητε, τα δικαιώματά τους ε, στη μητρότητα, προστασία των καταστάσει, βελτίωση τη συμμετοχή των γυναικών στην ε, ανοικοδόμηση μετά την εμπόλεμη σύραξη, την ανασυγκρότηση, πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις, πώς μπορούν να έχουν πολιτική συμμετοχή και τι ρόλο έχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Νομίζω ότι η κυρία Ματέρα ε, κινείται στις ίδιες γραμμές ε, σκέψης, το ίδιο μικρό με το σχέδιο γνωμοδότησής της. Θα καταθέσουμε λοιπόν και εμείς τροπολογίες μας. Σας είπα περίπου πώς για κατεύθυνση να κινηθούμε και φέτος υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ε, πηγαίνοντας και προς το 2015, οι, οποία, οι οποίες θα βοηθήσουν ε, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και την αύξηση των γνώσεων για το πώς θα καταπολεμηθεί και η άγνοια σε ό,τι αφορά την υπηρεξική βοήθεια ε, της Ένωσης, θα μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά για την βελτίωση της κατάστασης και σε τρίτες χώρες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόσωπος που θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τη γνωμοδότηση. Είναι πολύ χαροπιό για μα να βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την ανάπτυξη δεν αναπτύσσεται μόνο στην Επιτροπή Ανάπτυξη αλλά και εδώ. Το Ευρωπαϊκό Έτος της Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Έτος διοργανώθηκε τα τελευταία ε, χρόνια, 30 χρόνια και οργανώθηκε πρώτη φορά για θέματα που αφορούν εξωτερικές πτυχές πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα ευρωπαϊκά έτη είναι χρόνια που σχετίζονται με επικοινωνία, πρόθεση διαφόρων πτυχών πολιτικής. Γι' αυτό εδώ μιλάμε για την πρόθεση αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όλοι μας έχουμε επεξεργαστεί αυτό το θέμα επί μακρών. Και ο ρόλος των γυναικών και οι ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα των κοριτσιών να πάνε στο σχολείο είναι πράγματα που αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Συνένεση και στο πρόγραμμα για την αλλαγή και στο πλαίσιο μετά το 2015 που έχουν συγκεκριμένο κεφάλαιο για την ισότητα και τη δικαιοσύνη και την ισοτιμία και έχουμε και το σχέδιο δράσης 2014 την ισότητα των φύλων. Πριν από δύο χρόνια ο πρόεδρος Μπαρόζο δέσμευσε ένα δις ευρώ για πρωτοβουλίες σχετικές και για διάφορου φορεί που έμεναν πίσω και για τους στόχους της χιλιετίας. Και ένας από τους στόχους που έμενε πίσω ήταν η υγεία των μητέρων και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο θέμα και να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έχει χρηματοδοτήσει αυτούς τους στόχους και από το 2004 και μετά 7,5 εκατομμύρια γεννήσεις έγιναν στα, με τη βοήθεια ε, πολύ καλά κατατεσμένου προσωπικού και αυτό αύξανε τη δυνατότητα επιβίωσης και του νεογέννητου και των μητέρων. Λοιπόν, έχουμε τις ε, ημέρες τον επόμενο μήνα για την ανάπτυξη και θα έχουμε υψηλό επίπεδο, ένα πάνελ υψηλού επίπεδου για, που θα συζητήσει θέματα γυναικών και γυναικείων δικαιωμάτων και είναι στόχοι που θα προωθηθούν μετά το 2015. Έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε, το Ευρωπαϊκό Έτος της Ανάπτυξης και οι γυναίκες πράγματι θα εστιαστούν από αυτών των ζητημάτων. Τώρα κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος εμείς προσπαθούμε τους στόχους να τους έχουμε πολύ γενικούς και να μην εστιαζόμαστε σε μια συγκεκριμένη πτυχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα αν αυτό είναι και η άποψη του Κοινοβουλίου ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά εσάς και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την κυρία Παπαδοπούλου ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να καταπολεμήσουμε την άγνοια που υπάρχει όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Θα δώσω εκ νέου το λόγο στην κυρία Ρεζίνα Μπάστος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω, να την ευχαρίστησή μου για τα λόγια υποστήριξης και ευχαριστειών που ακούστηκαν όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Μπάρμπαρα Ματέρα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίδρασή της όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε τα διάφορα στοιχεία που έχουν αναφερθεί όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και τα στοιχεία δείχνουν ότι ε, σημαντικά ποσά, πολύ σημαντικά ποσά διατίθενται και διατίθενται σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα διαδοθεί το μήνυμα σχετικά με αυτά που κάνουμε σε αυτό το τομέα. Να το μάθουν οι πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους κυρίας Ματέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάστους. Και τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα εδώ στην Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναπτύξης θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του χρόνου τον Μάρτιο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και θα πρέπει να διακόψουμε για λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είχε προγραμματιστεί η ψηφοφορία για τις 10.45 και λάβαμε έτοιμα από την κυρία Μωράν Σαρτιέ που θα παρίσταται σε άλλη ψηφοφορία, σε άλλη επιτροπή και μας ζήτησε να εξετάσουμε την έκθεσή της λίγο πιο νωρίς. Θα της πω ότι τελειώσαμε νωρίτερα και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε 5 λεπτά, 5 λεπτά διάλειμμα. Vamos começar o nosso período de votação. Ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Um Πρώτη έκθεση που τίθεται σε ψηφοφορία είναι οι γυναίκες με αναπηρία. a relatora é a senhora Η συγκίτρια είναι η κυρία Βέρτμαν. Θέλετε κυρία Βέρτμαν να λάβετε το λόγο. Ευχαρίστω, αλλά στο τέλος παρακαλώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Επομένως να περάσουμε κατευθείαν στην ε, ψηφοφορία. Α, κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να πω εκ μέρους ε, της ομάδας του ΕΛΚΑ ότι τη ο σκιώδης για αυτή την ε, έκθεση ή μάλλον συνάδελφος Εστάρα, θέλει να αποσύρει το τροπολογία περιθυμών 1. Μάλιστα, πολύ ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβεβαστική 10, ψήφι υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 τροπολογία και 77 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 78, ψήφι Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 καταπίπτει. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Α, θα γίνει έλεγχος για την 113. Ξεκινά ο έλεγχος, η ψηφοφορία ηλεκτρονική, πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121. τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 15 υπέρ Το δεύτερο τμήμα μόνο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 126 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 10, πρώτο τμήμα κατά πίπτη. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Θα γίνει έλεγχος λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλοκτό υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 156. Τοπολογία 156 άρχεται η ψηφοφόρια. Πέρασε ψηφοφορία. Απερίφθη. Απασχόληση 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 αν ελέγξουμε την 178 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 178 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 187 υπέρ κατά αποχές ΔΒ DV3 υπέρ κατά αποχές ΔΒ DV4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δβ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. δβ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται.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 Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και θα ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Θέλει εισηγείται το λόγο. Η κυρία Βέρτμαν, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες τις σκιώδεις εισηγήτριες, καθώς επίσης τα μέλη της Γραμματείας για την θαυμάσια συνεργασία, επίσης για τις πολυάριθμες συμβιβαστικές τροπολογίες που μπορέσαμε να συντάξουμε για, ε, με βάση μια ε, συνεργασία ε, σε πλαίσιο σεβασμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας πάμε στην επόμενη ψηφοφορία για το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Η Πιτικάινεν Κάινεν Η κυρία Πιτικάινεν δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο, αν είναι εδώ. Όχι, εν τη αυτή περιπτώσει θα προχωρήσουμε και θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Συμβαστική 1. Υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπερκατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται προτιμώ να επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 9, ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 α όχι με συγχωρείτε πρώτα η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε επαληθεύσουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 Καλά, να επαληθεύσουμε λοιπόν την προηγούμενη. Νομίζω πάντως ότι παραμένει η ίδια πλειοψηφία. Αρχίζει η ψηφοφορία.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 Εγκρίνεται και αυτή. Τελική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. 17 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές και καμία, ε, συγγνώμη, 3 κατά, κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγητρία. Και προχωρούμε στην αμέσως επόμενη ψηφοφορία της γνωμοδοτήσεως. για θέματα ανάπτυξης του κράτους του Νότιου Σουδάν. Με εισηγήτρια την κυρία Τσέσκιοβα. Εσείς έχετε το λόγο τώρα κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα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 εγκρίνεται. Α, όλες μαζί λοιπόν ορισμένες τροπολογίες. 17 μέχρι τέλους. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία η οποία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλες. Πέρας. Υπέρ 19 ψήφι, ουδεμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια και πάλι στην εισηγήτρια. Και τώρα θα περάσουμε στο 10. Ψηφοφορία για την ηλεκτρονική υγεία για, την, για τον 21ο αιώνα καινοτόμος φροντίδα υγείας με εισηγείται την κυρία Ρονζούλη. Προχωρούμε αμέσως στην ψηφοφορία. Απολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε όμως. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, θέλετε από κοινού να τις ψηφίσουμε. Αντιρρήσεις υπάρχουν. Από την 8 λοιπόν 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, μέχρι το 14. Εντάξει, μέχρι εκεί. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται να ελέγξουμε όμως. Ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Τροπολογία 15, έτσι.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 19 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγητριά μας και περνάμε στο σημείο 11 της Μέσιας Διάταξης. Μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η συγχύτρια, μάλλον συντάκτρια της γνωμοδότησης, η κυρία Κορνέλισεν, η οποία απουσιάζει. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τρο, 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, ελέγχουμε, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. εγκρίνεται. 11 προς 7, τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ήταν η ίδια πλειοψηφία. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε καλύτερα την 59, άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 60 άρχη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και αυτή απορρίπτεται 61 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, Θα ελέγξουμε την 23. Απορρίπτεται κατά την άποψή μου, αλλά ελέγχουμε καλύτερα. Πέρας ψηφοφορίας. Πράγματι απορρίφθηκε. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 με μια προφορική τροπολογία υπέρ Α, ναι, υπάρχει πρώτα απ' όλα αντίρρηση προς την προφορική τροπολογία. Όχι, άρα τώρα ψηφίζουμε τροπολογία 66 με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 68 έχει αποσυρθεί. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, ελέγχουμε καλύτερα. Ελέγχουμε την 26, άρχη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 71 υπέρ. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, ελέγχουμε, ελέγχουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 29. Να ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβεβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33, καταπίπτει, όχι. Δεν καταπίπτει. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50, 36 ε, υπέρ κατά αποχές 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία τώρα. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της 41. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 40, ε, μάλλον 7 υπέρ. 7 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 44. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Ή κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει. Απορρίπτεται τέλος πάντων. Τροπολογή 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε την ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Ναι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 15 ψήφοι πέρα, 2 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε λοιπόν στην τελευταία ψηφοφορία. Όχι. Um, και που είναι η ψηφοφορία αφορά το Γενικό προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2014 όλοι οι τομείς. Προτείνω να ψηφίσουμε στο σύνολό του. Όχι. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οπότε εδώ ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα λάβει η χώρα στις 14 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι και θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών τώρα. Έληξε, διακόπτεται τη συνεδρία της Επιτροπής. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο για εκείνους που τελείωσε σήμερα η εβδομάδα τους. Και θα τα πούμε συνεδρίαση των συντονιστών, για τους συντονιστές που είναι παρόντες τώρα αυτό. Γεια σας.